Le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εστονίας, πρόεδρος Ήλβες. Liebe Kolleginnen und Kollegen, αγαπητοί αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι να εξαιρετική μου χαρά να χαιρετίζω τον κύριο Τόμας Ήλβε στο Κοινοβούλιο. Επέστρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς ήταν επί σειρά ετών Ευρωβουλευτής. Σήμερα έρχεται δεύτερη φορά ως πρόεδρος της Εστονίας. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ε, καλωσορίζω και σας δίνω και αμέσως τον λόγο. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της Εστονίας. Κυρίες και κύριοι, ζητώ συγγνώμη, η φωνή μου είναι βραχνιασμένη. Κάτι κόλλησα στην Εστονία. Πέρα από δέκα χρόνια έφυγα από αυτή την αίθουσα για να πάω στην ε, χώρα μου. Δεν υπήρχε μεταναστευτική κρίση, δεν υπήρχε ιδέα ότι μπορεί να αλλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα δια της βίας, ε, δεν έλεγε κανείς ότι μπορεί να αποτύχει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Δεν υπήρχαν έξυπνα τηλέφωνα, δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις από το ίντερνετ, δεν υπήρχε και Uber. Κυρίες και κύριοι, σχεδόν τα τρία τέταρτα ενός αιώνα επαναλαμβάνουμε το ότι η οικοδόμηση της Ευρώπης είναι για την ειρήνη. Για τρία τέταρτα ενός αιώνα, 75 χρόνια, η, Ευρώπη, η μισή Ευρώπη, για να ακριβολογούμε, κατάφερνε να ευημερεί παρά το ότι είχε αναθέσει σε κάποιους άλλους την ασφάλειά της, ακόμα και αν αντιμετώπιζε την Σοβιετική Ένωση. Απουσία λοιπόν εξωτερικών απειλών προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της Ευρώπης για να φέρουμε ε, εντός της Ευρώπης τις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονταν ε, υπό καταναγκαστικό καθεστώ. Σήμερα όμως αντιμετωπίζουμε νέες υπαρξιακές ε, απειλές και όπως μας υπενθυμίζει το Παρίσι και εσωτερικές απειλές η Ευρώπη πλέον για πολλούς δεν είναι η απάντηση. Εγώ ακούω τα λόγια του ποιητή, του Γέιτς στο ποιητή. Γυρίζοντας συνεχώς το γεράκι δεν μπορεί να ακούσει τον γερακάρι. Τα πράγματα διαλύονται και η ενέργεια χάνεται. Ας αντιμετωπίσουμε λοιπόν την νέα αυτή πραγματικότητα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κρίση μετασχηματισμού θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας ή θα το κάνουν άλλοι. Πρόκειται για μια κρίση η οποία θα δοκιμάσει ό,τι έχει επιτύχει η Ευρώπη βήμα-βήμα από την εποχή των Μονέ και Σουμάν. Φτάνουμε σε ένα σημείο κρίσιμο που είτε θα γίνουμε ισχυρότεροι είτε θα αφήσουμε τις φυγόκεντρες δυνάμεις να επικρατήσουν. Πρέπει να παραδεχτούμε πως σε αυτή την κρίση μετασχηματισμού πολλά πράγματα ήταν προβλέψιμα γνωρίζαμε πως υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, αλλά αναβάλαμε τις εσωτερικές κρίσεις ε, του ευρώ μέχρι να φτάσουν στο μη περαιτέρω την αντιμετώπιση τους ε, και θεωρούσαμε μέχρι πρώτον ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κάναμε λάθος. Γνωρίζαμε επίσης εδώ και καιρό πως οι τεράστιες διαφορές στο εισόδημα και τη δημοκρατία μεταξύ της Ευρώπης και της άμεσης γειτονιάς της ε, προς Ανατολάς και προς Νότον ήταν μια ορολογιακή βόμβα. Αλλά βεβαίως υπήρχαν κάποια απολυταρχικά καθεστώτα προς Νότον που συγκρατούσαν το ρεύμα στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η μαζική μετανάστευση και το ότι ο κόσμος φεύγει από τις σφαγές του εμφυλίου πολέμου και του Ισλαμικού κράτους μαζί με οικονομική μετανάστευση και φυγή από την φτώχεια απειλεί την Ευρώπη ως ποτέ άλλοτε. Η Σέγγεν απειλείται, κάποιες χώρες αρνούνται να δεχτούν πρόσφυγες, άλλες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια νούμερα. Η αλληλεγγύη καταραίει. Κάποιοι αρνούνται να βοηθήσουν, άλλοι δικαίως λένε πως η αλληλεγγύη είναι στη βάση της αμοιβαιότητας. Τα διαρθρωτικά ε, επίση κονδύλια είναι άλλη μια μορφή αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι, ακούμε εκπληκτικούς αριθμούς. Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ε, φέτος στην Ευρώπη και ε, προβλέψεις για άλλα δύο εκατομμύρια αυτό το έτος. Ναι, είναι μεγάλη αριθμή, ναι, θα δοκιμάσουν την κοινωνική συνοχή, τον προϋπολογισμό και όμως έχουμε δει πολύ χειρότερα και έχουμε επικρατήσει. Στην Ευρώπη του 1946 στη Γερμανία μόνο υπήρχαν 12 εκατομμύρια εσωτερικοί πρόσφυγες και άλλα 12 εκατομμύρια ε, εκτοπισμένοι από 20 διαφορετικές χώρες. Για να επιληθεί αυτό η Ούνρα, η υπηρεσία του ΟΗΕ, εξόδεψε αυτό το οποίο σήμερα αναλογεί σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρω αυτό το νούμερο για να έχουμε μία ιδέα του πόσο τεράστια ήταν αυτά τα οποία αντιμετώπιζαν ε, οι παππούδες μας όταν η Ευρώπη δεν είχε αχιαπλαθισμούς αλλά ούτε καν κυρίαρχα κράτη. Και όλα αυτά πριν ξεκινήσει καν το σχέδιο Μάρσαλ. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ας ε, ξεκινήσουμε τώρα ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας σταματήσουμε να δείχνουμε ο ένας τον άλλον με το δάχτυλο, θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση εάν επιδείξουμε την αποφασιστικότητα των προγόνων μας. Πρέπει να στάθουμε στο πλευρό των κρατών μελών που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος, πρέπει να δοθεί μια μορφή να το μοιραστούμε. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε πλήρως τα εξωτερικά σύνορα της Ένωση. Δεν μπορεί να, έχουμε, να μην έχουμε σύνορα ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Μα δεν θα τελειώσω έτσι. Πρέπει να υπάρχει και μια κοινή πολιτική ασύλου ειδικά όσον αφορά την απόρριψη προφανώς αστήρικτων ετοιμάτων και τον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών. Είναι τόσο δύσκολο αν σκεφτούμε το τι κάναμε τα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Κυρίες και κύριοι, μετά τις επιθέσεις του Παρισιού φοβάμαι πως ε, η κρίση αυτή των ε, προσφύγων θα οδηγήσει σε άνοδο λαϊκιστών και εξτρεμιστών. Θα δούμε το επιχείρημα, το είδαμε δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τους πρόσφυγες γιατί είναι τρομοκράτες, ξεχνώντας ε, πως αυτοί οι οποίοι σειραίουν σήμερα στην Ευρώπη φεύγουν από το ίδιο καθεστώς το δολοφονικό που είδαμε στο Παρίσι αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ο πολιτικός λόγος σήμερα υιοθετεί γλώσσα που πριν από λίγα χρόνια ε, ήταν σε ανώνυμα φόρα online. Κεντρώοι δημοκράτες ε, ηγέτες ε, δέχονται όλο και περισσότερες πιέσεις, να μην πω επιθέσεις. Τα ακραία κόμματα και οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται την κρίση αυτή όπως εκμεταλλεύτηκαν και την οικονομική κρίση, εκμεταλλεύονται την δυσαρέσκεια των φορολογουμένων με το να αναδεικνύουν την χλιαρή αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών. Όταν τα παραδοσιακά κόμματα λοιπόν δεν παρέχουν λύσεις, οι πολίτες στρέφονται σε αυτούς των οποίων η ρητορία ακούγεται αποφασιστική, αλλά είναι συχνά απλές και μη ευρωπαϊκές λύσεις. Η Ένωση δημιουργήθηκε ακριβώς για να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λέω μεταξύ άλλων ως ιός προσφύγων που έφυγαν από την χώρα μας, στην Εστονία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Γι' αυτό έχω αυτή την προφορά. Οι γονεί μου δεν αισθάνονταν πάντα καλοδεχούμενοι όταν έφτασαν στην Σουηδία αλλά τους δόθηκε μια ευκαιρία και ελπίζω σε λίγες δεκαετίες από σήμερα να υπάρχει ένας ε, πρόεδρος μιας δημοκρατικής Συρίας που θα μιλάει αραβικά με γερμανική προφορά. Κυρίες και κύριοι, έπρεπε να έχουμε προβλέψει την κρίση του ευρώ και της μετανάστευσης. Αυτό το οποίο δεν προβλέψαμε και πραγματικά είναι αδιανόητο είναι η εισβολή και η προσάρτηση της Κρυμαίας και η εισβολή στο Ντονμπάς. Δεν θα επιμείνω. Απλά θα πω πως με το να κάνει αυτό το οποίο έκανε πριν από δύο χρόνια η Ρωσία παραβίασε κάθε ευρωπαϊκή συνθήκη ασφαλείας. Ξεκινώντας από τη Χάρτα Ασφαλείας του ΟΗΕ την τελική πράξη του Ελσίνκη του 1975 και την Χάρτα των Παρισίων του 1990 και παραβίασε και την, το υπόμνημα της ε, Βουδαπέστης ε, του 1994 στο, το οποίο εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα να παραδώσει η Ουκρανία το τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό πλωστάσιο στον κόσμο που είχε τότε. Εν ολίγης, στην Ευρώπη δεν μπορούμε πλέον να υποθέτουμε ότι οι συνθήκες που εγγυώνται την ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή λέγω ασφάλεια από τον δεύτερο παγκόσμιο εξακολουθούν να ισχύουν. Οι είπα ήταν γρήγορες στην αντίδρασή τους και ο ΙΕ και αυτό βεβαίως είχε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις κυρώσεις. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με διαφορετική προσέγγιση της λεγόμενης στρατηγικής υπομονής. Κάποιοι λένε διάλογος. Ναι, ο διάλογος δεν είναι πολιτική και οπωσδήποτε δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε μάθει από το Μόναχο το 1938. Κυρίες και κύριοι, μίλησα για ευρωπαϊκές κρίσεις, κάποιες έπρεπε να έχουμε προβλέψει, άλλες όχι. Τώρα θα αναφερθώ στο μέλλον μας. Και σε μακροπρόθεσμη κρίση που μπορούμε να αποφύγουμε αν την πάρουμε στα σοβαρά πριν βρεθούμε εν το μέσο της. Η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της Ευρώπης μειώνεται σε έναν κόσμο ο οποίος διασυνδέεται. Μαζί με τον ε, κύριο Μπασού, τον ε, επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, ολοκληρώσαμε την μεγαλύτερη μελέτη για το οικονομικό δυναμικό της πληροφορικής και τη βελτίωση της ε, κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Επίσης αναδεικνύονται οι κίνδυνοι του να μείνει κανείς πίσω. Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη τα πάει καλά στην μελέτη αυτή που μας πήρε 1,5 χρόνο, αλλά να είστε σίγουροι η Ευρώπη θα γίνει δύναμη δεύτερης κατηγορίας καθώς όχι μόνο η ΙΠΑ αλλά η Ινδία και η Κίνα θα αναλάβουν ηγετικέ θέσεις εάν δεν κάνουμε τίποτα. Η ψηφιακή επανάσταση θα μπορούσε να βοηθήσει την ενιαία αγορά. Σήμερα βλέπουμε πανευρωπαϊκές αγορές ε, εν τη γενέση τους ε, στον τομέα της υγείας, μεταφορών και τραπεζών που πριν από λίγα χρόνια ήταν τελείως τοπικές αγορές αλλά η νομοθεσία μας παραμένει κατακαιρματισμένη μεταξύ κρατών μελών και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για την ψηφιακή εποχή. Χάνουμε γιατί δεν υπάρχει ενιαία αγορά, οι καλύτεροι και εξυπνότεροι φεύγουν εκεί όπου υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτό το είδα με τα ίδια μου τα μάτια όταν ένας 23χρονος ε, βρήκε λίγα χρήματα και τον είχα προσκαλέσει ε, να με συναντήσει και μου είπε κύριε πρόεδρε φεύγω πάω στη ΣΥΠΑ. Του λέω γιατί μου λέει εκείνη οι ευκαιρίες. Μετά από έξι μήνες είχε, είχαν επενδύσει στην εταιρεία του 4,5 εκατομμύρια δολάρια και τρία χρόνια μετά την πούλησε για 100 εκατομμύρια δολάρια. Μπορούσε να είχε μείνει στην Εστονία αν είχαμε ενιαία αγορά και υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση. Και μπορώ να σας αναφέρω τέτοιες ιστορίες από όλες τις χώρες της Ένωσης. Πριν από 60 χρόνια όταν η συνθήκη της Ρώμης έθεσε τις βάσεις των τεσσάρων ελευθεριών, ελεύθερη διακίνηση προσώπων αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, δεν υπήρχε ψηφιακά τίποτα. Υπολογιστές δεν υπήρχαν. Σήμερα μιλάμε σε ένα, ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Εάν δεν αναγνωρίσουμε πόσο Βαθιές είναι αυτές οι αλλαγές, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Η Ευρώπη θα μείνει πίσω και οι πολίτες μας το ίδιο. Το να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ψηφιακής επανάστασης σημαίνει πως θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι επιχειρήσεις της Ευρώπης, η κοινωνία των πολιτών και τα κράτη. Οι δυνάμεις της αγοράς ε, και τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στην αλλαγή, αλλά η νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να τις στηρίξει. Για να δούμε το μέγεθος της αλλαγής προτείνω να προσθέσουμε στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες μία πέμπτη ελεύθερη διακίνηση δεδομένων. Η πέμπτη αυτή ελευθερία μπορεί να ενταχθεί ε, θα έλεγε κανείς τις ε, τέσσερις προηγούμενες αλλά σήμερα πλέον νομίζω πως είναι διακριτή και πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά τα δεδομένα δεν είναι ούτε πρόσωπο, ούτε υλικό αγαθό, ούτε κεφάλαιο, ούτε υπηρεσία. Αλλά πρέπει και τα δεδομένα να μπορούν να κινούνται διασυνοριακά. Η πρόταση της Κομισιόν για ενιαία ψηφιακή αγορά ακριβώς ε, θα θέσει τα θεμέλια της ελευθερίας δεδομένων, αλλά θα πρέπει να είναι θεμέλιο τη κοινή αγορά, όχι ένα στόχο που πρέπει να επιτευχθεί. Από την πλευρά των πολιτών, τι θα σημαίνει η πέμπτη ελευθερία. Πρώτα απ' όλα, ελεύθερη διακίνηση δεδομένων σημαίνει πω θα έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίε που πληρώνουμε σε ολόκληρη την Ένωση. Σημαίνει πω το εμπόριο στο διαδίκτυο δεν θα περιορίζεται από τη χώρα που έχουμε τραπεζικό λογαριασμό και τα εθνικά σύνορα δεν θα καθορίζουν ε, ποιοι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να αγοράσουν ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες και ποιοι όχι. Οπότε σήμερα ε, είναι ευκολότερο να στείλουμε ένα μπουκάλι ελαιόλαδο από τη Σικελία στο ναρκτικό κύκλο από ότι ένα τραγούδι στο iTunes ε, από τη μια χώρα στην άλλη. Και καθώς ε, φυσάω τη μύτη μου να σας πω πως στην χώρα μας οι συνταγές, οι ιατρικές είναι ψηφιακές. Οπότε ο γιατρός μου μπορεί να μου γράψει μια συνταγή και να πάω σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Αλλά αυτό δεν γίνεται εκτός Εστονίας και δεν βλέπω το λόγο γιατί. Γιατί να πάω σε ένα φαρμακείο εδώ στο Ρασβούργο και να πάρω το φάρμακο που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή με μια συνταγή που θα μου γράψει ο γιατρός μου στην Εστονία είναι εφικτό, δεν υπάρχει τεχνολογικό πρόβλημα και στην νομοθεσία μας υπάρχει. Όμως η ελεύθερη διακίνηση δεδομένων δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Όπως και οι άλλες θεμελιώδεις ε, ελευθερίες ε, φέρνει μαζί της ευθύνες, ε, δικαιώματα δηλαδή και υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Και βεβαίως αυτό σημαίνει προστασία των δεδομένων. Το να έχει κανείς ε, έλεγχο των δεδομένων του είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ακριβώς την αξία αυτών των δεδομένων. Ο νέος γύρος λοιπόν ε, διαπραγματεύσεων και σας συγχαίρω για αυτό το οποίο κάνατε ότι ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις αναγνωρίζει το πράγμα αυτό επί της ουσίας και θα έχουν πραγματικά έλεγχο επί των δεδομένων τους οι ενδιαφερόμενοι θα δημιουργηθούν έτσι νέες αγορές και θα μειωθεί η χαρτούρα και η γραφειοκρατία του δημοσίου τομέα που κοστίζει αυτή τη στιγμή στους πολίτες ε, απογοήτευση και χρόνο και χρήμα και θα αυξήσει δραματικά την διαφάνεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια οικονομία των δεδομένων και για μη προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αξία που κρύβεται στα μεγάλα δεδομένα, όπως λέγεται, που δημιουργούν τα ηλεκτρονικά μας αυτοκίνητα, σπίτια, ψυγεία ή συνδεδεμένες αυτές συσκευές. Αυτό το οποίο στη Γερμανία ήδη σήμερα ονομάζουμε βιομηχανία 4.0. 4,0. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να δημιουργήσει ακριβώς την ασφάλεια αυτή που θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη, ειδικά η τεχνολογία blockchain η οποία θα προωθήσει πάρα πολύ την χρήση Τέλος χρειαζόμαστε βεβαίως όπως χρειαζόμαστε για την διακίνηση αγαθών, δρόμους και λιμάνια χρειαζόμαστε και εδώ πέρα την απαραίτητη υποδομή. Οι συνδέσεις ε, πέμπτης γενιάς, οι οπτικές σύνες πρέπει να φτάσουν πραγματικά παντού στην Ευρώπη, στο λεγόμενο τελευταίο χιλιόμετρο, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Οι περιοχές υπαίθρου που έχουν αποφεληθεί τόσο πολύ από την κοινή γεωργική πολιτική απαιτούν στον νέο αυτόν κόσμο την ίδια πρόσβαση στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον στην πόλη. πρέπει επίσης τα ωφέλη του ψηφιακού αυτού μερίσματος ε, να τα απολαμβάνουν όλοι. Η εμπειρία της Εστονίας τουλάχιστον με καθιστά αισιόδοξο από το 2005 επιτρέψαμε την ψηφοφορία στο διαδίκτυο σε νέα τοπικές, εθνικές ε, και δημοτικές εκλογές. Μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό αφορά τους νέους των πόλεων που είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Όμως οι μελέτες δείχνουν ξανά και ξανά πως δεν υπάρχει χάσμα είτε δημογραφικό είτε αστικό και της υπαίθρου. Ο συνταξιούχος της υπαίθρου ψηφίζει ε, όσο και ο νέος πόλης μιλάει ε, στο Skype με την οικογένειά της ε, και ανέφερα το Skype βεβαίω γιατί επρόκειτο για εστονική εφεύρεση αλλά όπως και πολλά άλλα πράγματα πλέον βρίσκεται στο Redmond της, Washington, της πολιτείας Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα πρέπει να ρωτήσουμε πού μας πηγαίνει αυτή η ψηφιακή επανάσταση, ποιο είναι το μέλλον της εργασίας στην ε, ψηφιακή εποχή, τι θα συμβεί στη δουλειά του βιομηχανικού εργάτη και του ταξιτζή. Και αύριο μεθαύριο στη δουλειά του γιατρού και του λογιστή. Κάθε προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση αύξησε την απασχόληση αντικαθιστώντα παλιέ δουλειέ με καινούργιες που απαιτούσαν περισσότερε δεξιότητε και πλήρωναν περισσότερο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει το ίδιο και τώρα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της ψηφιακής επανάστασης και εγώ έχω την ταπεινότητα να παραδεχτώ πως δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Αλλά γνωρίζω το εξής. Η ψηφιακή επανάσταση όπως και η κρίση της Ευρωζώνης, της Κρυμαίας και των προσφύγων απαιτούν από εμά να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας τη στιγμή που η πολιτική απευθύνεται στα πιο χαμηλά ένστικτα να μην υποθέτουμε πως είναι ε, κρίσεις που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα των προκατόχων μας. Το 1957, το 1989, το 1991 και το 2004. Και αυτοί αντιμετώπιζαν αβεβαιότητα αλλά προχώρησαν. Εάν υποκύψιμους λαϊκιστές που λένε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το συμφέρον των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε καμία κρίση προβλέψιμη ημί δεν θα αντιμετωπιστεί την μετανάστευση, το ευρώ, ακόμα και στρατιωτικές επιθέσεις, να μην αναφέρω την πρόκληση της τεχνολογικής αλλαγής καν. Οι λύσεις οι οποίες μας επαναφέρουν στο έθνος κράτος θα μας φέρουν σε μια κατάσταση πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου θα σκεφτόμαστε πώς θα βλάψουμε τον γείτονα και βεβαίως ε, θα πάμε στο οφθαλμόν αντιοφθαλμού. Σε μια εποχή όπου ξανά θα ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Και έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της Ευρώπης που οδηγεί αυτό. Ας μην έχουμε ψευδεστήσεις για το τι θα γίνει εάν διστάσουμε. Γιατί, όπως είχε πει ο Γέιτς, στο ίδιο ποίημα, η καλύτεροι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ενώ οι χειρότεροι είναι απολύτως σίγουροι για το τι θέλουν. Η επιλογή είναι δική μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα λόγια που είπατε δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Νομίζω το χειροκρότημα και οι διαμαρτυρίες ε, μιλάνε από μόνα τους. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κύριος Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ πάρτε τις θέσεις σας. Ε, η κυρία Άτκινσον έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας. Κυρία Άτκινσον, ποιο είναι το θέμα επί της διαδικασίας. Παρακαλώ, αναφερθείτε στο θέμα επί της διαδικασίας. Είναι νομικό θέμα που συνέβη στην χώρα μου, που θεωρώ πως αφορά το σώμα. Απαλλάχθηκα από όλες τις κατηγορίες ε, ε, που υπήρχαν εναντίον μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που με στήριξαν. Από όλες τις ε,